Καλημέρα σε όλους σας αγαπητοί φίλοι. Θα ξεκινήσουμε. Θα μιλήσω ισπανικά. Λοιπόν, αν χρειάζεται μετάφραση να τα ακουστικά σας. Antes Πριν ξεκινήσουμε την εξέταση της ημερήσιας διάταξης της σημερινής μας συνεδρίασης, θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι και να σας πω κάτι. Χθες στην Ισπανία, πέντε άνθρωποι, πέντε αθώοι, τρεις γυναίκες και δύο παιδιά δολοφονήθηκαν. Είναι αυτό από το κος του ματσίσμου της βίας λόγω φίλου. Δυστυχώς ε, δεν είναι στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων ευρωπαϊκών εφημερίδων αυτό αλλά μιλούμε και για τρομοκρατική πράξη. Πέντε άνθρωποι σε μία μόνο μέρα, σε μία μόνο χώρα. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα θύματα της βίας φίλου, λόγω του φίλου και αλλού στην Ευρώπη, όμως αξίζει να εκφράσουμε το σεβασμό μας στα θύματα και στις οικογένειές τους και γι' αυτό ζητώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Muchas Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην λησμονούμε ποτέ την ευθύνη που έχουμε όλοι μαζί και ο κάθε ένας από μας ξεχωριστά. Για τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να τελειώσει πια αυτή η κοινωνική βαρβαρότητα. Περνούμε στην εξέταση της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις του Προέδρου. Ως προς την ε, προετοιμασία του προϋπολογισμού 2016 πρέπει να καθορίσουμε τις εκάστοτε ομάδες για τις πιλωτικές δράσεις και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και γι' αυτό η Γραμματεία θα έρθει σε επαφή με τις πολιτικές ομάδες για να τις ενημερώσει για το περιεχόμενο, για τη διαδικασία και για να μπορέσουν οι πολιτικές ομάδες να συμβάλλουν σε αυτό το εγχείρημα. Επίσης, στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών που έλαβε χώρα αμέσως πριν, ενέκριναν οι συντονιστές την εκπόνηση των εκθέσεων που θα συντάξει η Επιτροπή μας, όρισαν τους εισηγητές και τις εισηγήτριες, και αποφάσισαν για τις ακροάσεις και τις ε, διοργανώσεις των ακροάσεων για τη φετινή χρονιά, καθώς και για τις προτάσεις διοργάνωσης αποστολών. Και ο συντονιστής της εκάστοτε πολιτικής ομάδας θα ενημερώσει τους ε, συναδέλφους και τι συναδέλφους. Περνούμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ψήφιση των εκθέσεων. Αν έχετε τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας μπορούμε να ξεκινήσουμε. Η κυρία Μορβάη θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάνω λάθος. Θεωρώ όμως ότι σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να συνοψίσετε την συνεδρίαση των συντονιστών. Τι αποφάσεις να μας ενημερώσετε. Με ενδιαφέρει. Διότι με μια γεγραμμένη και κανονικά εξαιρούμε από την ε, ενημέρωση. Αν δεν κάνω λάθος, ο κανονισμός απαιτεί να το κάνετε αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ αν μπορείτε να αποκαλύψετε τι αποφασίστηκε συνεδρία των συντονιστών. Ε, ναι, κυρία Μορβάη θα πάρετε εσείς τις πληροφορίες, θα σας τις στείλουμε ακριβώς όπως θα το διαβιβάσουμε και στις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Σε είπα ήδη ότι οι συντονιστές έλαβαν αποφάσεις για το ποιες εκθέσεις θα καταρτήσει η Επιτροπή μας, για το ποιοι θα είναι οι συγητές που θα συντάξουν τις εκθέσεις αυτές, για το ποιες ακροάσεις θα οργανωθούν, καθώς και το ποιες αποστολές θα οργανωθούν κατά τη διάρκεια του 2015 και εξέτασαν και δύο προφορικές ερωτήσεις που θα τεθούν προς συζήτηση στην Ολομέλεια και για μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή θα σταλεί το περιεχόμενο των προφορικών ερωτήσεων στους συναδέλφους για να μπορούν να τις μελετήσουν, να παρουσιάσουν τροπολογίες. Και αυτό θα γίνει στην συνεδρίαση της Επιτροπής 5 και 6 Μαΐου. Εκεί θα εγκρίνουμε το περιεχόμενο των προφορικών ερωτήσεων. Και εσείς προσωπικά θα λάβετε όλα αυτά τα στοιχεία και όλες αυτές τις πληροφορίες. Περνούμε τώρα, όπως έλεγα, στην ψήφιση των εκθέσεων. Καταρχάς έχουμε την έκθεση για την ανάπτυξη και την απασχόληση, προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση. Ξεκινούμε με τη συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 τροπολογία υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Θέλετε να υπαλθεύσουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 31. Ψηφίζουμε τώρα δια της ηλεκτρονικής οδού την τροπολογία 31. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 32. Ψηφίζουμε την 32 έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Είμαι σίγουρη ότι η Προεδρία μπορεί και να κάνει λάθος, αλλά βλέπω ότι όταν υπάρχουν περίπου τα ίδια χέρια σηκωμένα, ο ίδιος αριθμός πάνω κάτω από τη μία και από την άλλη μεριά, τότε επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Και αν εσείς θέλετε οποιαδήποτε στιγμή να το επαληθεύσουμε, παρακαλώ να το πείτε. 33 τροπολογία, σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν έχουμε ψηφίσει 34. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Στον κατάλογο ψηφοφορίας έχω σημειωμένο ότι την 33 και την ψηφοφορία κατά τμήματα ζητά το ΕΛΚ. Και άρα πρέπει να την ψηφίσουμε κατά τμήματα. Αυτό έχω σημειώσει. Καλώς. Το πρώτο τμήμα της 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26. Όχι, συγγνώμη. Η 41. Τροπολογία 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές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 αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Ψηφίζουμε την τροπολογία 53 δια της ηλεκτρονικής οδού. Πέρας της ψηφοφορίας. Καλά το είχα δει. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ. 11 κατά. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ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 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις, τα εκτιμώντας. Έχετε προφορική τροπολογία, παρακαλώ. Έχω, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν μπούμε στις αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 3, αιτιολογική σκέψη α, της κυρίας Μπιλμπάου, με δική της συμφωνία από ό,τι καταλαβαίνω μπορώ να πω ότι θα πρέπει να λέει. Εκτιμώντας ότι ιστορικά οι γυναίκες επλήγονται περισσότερο από την ανεργία από ότι άντρες, εκτιμώντας ότι την ενεργία των γυναικών στο 10% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικές διαφοροποίησεις και ο στόχος για έχοντας σαν στόχο να διαπιστώσουμε ότι η οικονομική κατάσταση των γυναικών έχει επιδεινωθεί από όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση. Si Εάν συμφωνούμε όλοι, ψηφίζουμε με το... να συμπεριληφθεί αυτό στο κείμενο. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Ε, ψηφίζουμε την τροπολογία επαριθμών 1. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9. Τροπολογία. Υπέρ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 Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το επαρθέσουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Ψηφίζουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία όλη τη έκθεση. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Ομόφωνα. Συγχαρητήρια, κυρία Γκέρλιν. Εγκρίνεται η έκθεσή σας. Pasamos al Περνούμε στην, κατάσταση, στην έκθεση σχετική με την πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Κυρία Λεγκρίπ, θέλετε το λόγο. Ναι, στα γρήγορα, διότι η συγγήτριά μας η κυρία Γκάμπριελ δεν μπορεί να παρίσταται εδώ και με επιφόρτησε με το να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου τη, γιατί επιστρέφει στην πατρίδα τη. Ευχαριστεί εκ βάθου καρδία όλε τι συνηγήτριε και όλου του συναδέλφου που κατέθεσαν ανθρωπολογίε. Οι περισσότερε θα στηριχθούν και θα εμπλουτίσουν το σχέδιο γνωμοδοτήσεω. Κύριε Γκαμπριέλ, θέλω να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών ότι, σαν αναπληρωματικό μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μα, θα εργαστεί ούτω ώστε οι συστάσει τη Επιτροπή Γυναικών να ληφθούν επαρκώς υπόψη και να σωματωθούν τη στιγμή της ψηφοφορίας ε, στο κείμενο που θα, το οποίο θα επιληφθεί η Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ η κυρία Μπεσέρα. Ναι κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εάν είναι δυνατό θα ήθελα να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία η οποία θεωρώ ότι εμπλουτίζει αυτή την πρωτοβουλία που αναφέρεται σε αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί πρόσφατα. Εκτιμώντας ότι ε, στις 19 Μαρτίου χτυπήθηκε μέχρι θανάτου η συγκεκριμένη γυναίκα αυτό δείχνει την τρομακτική πραγματικότητα των γυναικών στο Αφγανιστάν. Δηλαδή θέλουμε την προφορική τροπολογία να δείξουμε ε, τη βαρβαρότητα των κατηγοριών, να δώσουμε ονοματεπώνυμο σε αυτό. Ήταν η ομάδα γυναικών που κουβάλησε το φέρετρο αυτής της ε, γυναίκες και νομίζω ότι θα αποτίσουμε καλύτερο φορό τιμής έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Πεθέρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. θα το ψηφίσουμε και η γραμματεία θα δει σε ποιο σημείο του κειμένου ταιριάζει περισσότερο. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμό 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 4. Α, συγγνώμη, το έχουμε ψηφίσει. Την 6, συμβιβαστική τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7, συμβιβαστική 7, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές δεν το έχω σαφές στο μυαλό μου ψηφίζουμε την τροπολογία 29 δια της ηλεκτρονικής οδού πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Μαζί με την προφορική τροπολογία που μπήκε στο κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 33, απορρίπτεται 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Περνούμε στις ιδεολογικές σκέψεις. Θα ψηφίσουμε πρώτα την προφορική τροπολογία της κυρίας Μπεθέρα. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και περνούμε στην τροπολογία παριθμών 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Με προφορική τροπολογία μαζί, η οποία προσθέθηκε στο κείμενο. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το τελικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 29 ψήφοι υπέρ και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Γκάμπριελ. Περνούμε τώρα στην ψήφιση της έκθεσης για το ReFit. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Τροπολογία σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη ψήφιση της τελευταίας έκθεσης της κυρίας Σίλβια Κώστα. Τροπολογίες για το gender mainstreaming. Παράγραφος 17. Τροπολογία 2, ή μάλλον σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και η τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ψηφοφορία τη σημερινή. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Αν έχει την καλοσύνη, καθίστε. Um, Uh, I will speak uh, Θα μιλήσω πορτογαλικά. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας και τη συζήτησή μας. Η συζήτησή μας αφορά μια έκθεση που επεξεργάζεται από καιρό η Επιτροπή μας και αφορά την αφορμογή της οδηγίας 2006 κάθετος 54 περί της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας και της αντιμετώπισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία. Η κυρία Ζαμπόσκα είναι η συγγήτρια. Πριν αναφερθούμε όμως στην ε, γνωμοδότηση, συγκεκριμένο κείμενο, θα συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονές μας που παρίστανται εδώ σήμερα το πρωί, οι οποίοι θα μας δώσουν σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την έκθεση. ασχολούμεθα με θέματα που άπτονται της εφαρμογής της οδηγίας. Έχει, έχει, έχει γίνει κάποια απόπειρα από την ομάδα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η οδηγία και σήμερα το πόρισμα της μελέτης που ε, ανετέθη στην Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι κάτι που θα μας γνωστοποιηθεί. Ότως ώστε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ζώσεφ Ντάν που είναι διευθυντής της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολείται με την αξιολόγηση συνεπειών και την ευρωπαϊκή υποστηθέμενη αξία. Ο κύριος Ντάν λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικότατος, θα ήθελα να αναφέρω ότι στη Γενική Διεύθυνση της Υπηρεσίας της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έρευνα προσπαθούμε να στηρίξουμε την έκθεση της κυρίας Ζαμπόρσκα και αυτό στα πλαίσια της στήριξης των επιτροπών και του ελέγχου αξιολόγησης συνεπειών για τις εκθέσεις τις νομοθετικές ιδίας πρωτοβουλίας και τις διάφορες εκθέσεις. Γι' αυτό δημιουργηθήκαμε σαν φορέας. Στατηγική μας η πολλαπλή εισρωή πληροφοριών από τους εμπειρογνώμονες για να μπορούμε να βοηθούμε την Επιτροπή και να στηρίζουμε και την εισηγήτρια και τους ηγητές. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλώ στην Επιτροπή σας. Έγινε πολύ σημαντική εργασία πολιτική της Επιτροπής στην προηγούμενη θητεία και να επενθυμίσουμε ότι ετοιμάσαμε μια έκθεση που αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, στηρίζοντα την κυρία Μπάουερ που είχε ασχοληθεί με το ίδιο θέμα. Είναι έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας νομοθετικού περιεχομένου που ετοιμάστηκε στην προηγούμενη θητεία και αν δεν σφάλω, η κυρία Ζαμπόσκα ήταν η δεύτερη ε, η κυρία Ζαμπόσκα ασχολείται με δεύτερη τρίτη με αυτό το θέμα. Έχουν γίνει και άλλες απόπειρε, θα θυμόσαστε την ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά αυτή την έκθεση ε, ιδίας πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου. Ήταν πολύ απογοητευτική η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χώρισε και είναι συνετό αυτό που έκανε η Επιτροπή και εξετάζει με πρωτοπόρο τρόπο ε, την προσέγγιση από διάφορες οπτικές γωνίες. Ελπίζω να σας δώσει οπτικές γωνίες. Η ο Δόκτωρ Μπούρη θα δώσει ενδιαφέρουσα οπτική όσον αφορά την ενσωμάτωση του εθνικό δίκαιο, διότι η εφαρμογή από τρία μέρη, ενσωμάτωση του εθνικό δίκαιο, εφαρμογή, επιβολή και υλοποίηση. Από όλε τι εκθέσει λοιπόν θα δείτε διάφορες πτυχές που ήδη αναφέρονται σε πρώτες εργασίε Επιτροπής όπως ο ρόλος των φορέων περισσότητας, τα προβλήματα με τη συλλογή στοιχείων στα κράτη-μέλη και ούτω καθεξής. Θα αφήσω βέβαια τους εμπειρογνώμονες να τοποθετηθούν από αυτού. Νομίζω ότι είναι το πολιτικό ζήτημα που ελπίζουμε να οδηγήσει σε περαιτέρω εργασίες ε, και περαιτέρω ε, τοποθετήσεις και εργασίες από πλευρά της Επιτροπής. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ντάν. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον πρώτο αγορητή και είναι η καθηγητής ε, καθηγήτρια Σουζάν Μπούρη, με ο, η οποία είναι λέκτορ στη νομική σχολή της Ουτρέχτης και συντονίστρια στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπορογνωμόνων στον τομέα της ισότητας των φύλων, μπορεί να αναλύσει την εφαρμογή της οδηγίας εξετάζοντας εν γέννη τις νομικές πτυχές και πιο συγκεκριμένα την οδηγία περί διακρίσεως. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Σε αυτή την ε, συζήτηση έχουμε νέο ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμένων, όχι μόνο για την ισότητα των φύλων και για την αποφυγή των διακρίσεων και με ειδική ε, συντονίστρια για την ισότητα των φύλων. Ετοίμασα ένα έγγραφο που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας αναδιατύπωσης Ίρικας της οδηγίας εστιάζεται επί των ενιών της άμεσης και της έμεσης διακρίσεως κάλυψα ευρύτερο πεδίο κάπως, δηλαδή προέβην σε νομική ανάλυση της ε, οδηγίας για την αναδιατύπωση των κειμένων, ασχολούμαι τις βασικές ε, διατάξεις οδηγίας και την ομολογία τη σχετική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επιπλέον, Υπάρχει και ενδελεχής ανάλυση που αφορά έξι κράτη-μέλη. Έχει δημιουργηθεί ανάλυση. Οι εθνικοί εμπορογνώμονε απάντησαν σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο επ' αυτού. Νομίζω ότι ω νομικός πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το εξή. Η δευτερογενής νομοθεσία που συμπεριλαμβάνει στην οδηγία δεν μπορεί να, να, μετα... να τροποποιήσει τον πρωτογενή ε, την πρωτογενή νομοθεσία όπως ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης ε, αξίας. Αλλά μπορεί να δώσει εξηγήσει. Η οδηγία εν αυτή τη ενία έχει σημαντικό ρόλο. Σημαντική πτυχή είναι και η εξή. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των διαφόρων νομοθεσιών και οδηγιών για ισότητα των φύλων και αποφυγής διακρίσεων. Παραδείγματο χάρη οι ορισμοί και οι οριζόντιες διατάξεις πρέπει να συντονίζονται, όπως το βάρος της απόδειξης, η επιβολή κυρώσεων. Νομίζω είναι εξίσου σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την σχετικότητα του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθήκων ιδιαίτερος των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Καμιά φορά η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν είναι πολύ συνεπής και δεν συνάδει με κάποιες διατάξεις που είναι σχετικές για το θέμα και που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη παραγματος χάρη σχετικά με τη θετική δράση για τις γυναίκες. Η οδηγία περί ενδιατυπώσεως, recast, αφορούσε αναδιατύπωση του, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γίνεται εξίσου μια αναδιατύπωση του εθνικού δικαίου, ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Σε κάποια κράτη-μέλη ε, νέα νομοθεσία έχει εγκριθεί, όμως σε άλλες χώρες δεν θεωρήθη αναγκαίο κάτι τέτοιο για την εφαρμογή της οδηγίας. Συζητώ στο έγγραφό μου δύο επιλογές. Η πρώτη. Έχουμε σαν στόχο μια νέα οδηγία και η έκθεση της κυρίας Μπαόρ και το σχέδιο εκθέσεως της κυρίας Ζαμπόρσκα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια νομοθετική πρόταση για την αντικατάσταση της οδηγίας. Κατά την άποψή μου, μια νέα οδηγία θα επέφερε κάποια ωφέλη και κάποια μειονεκτήματα. Θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά τα στοιχεία. Πρώτον, θα αποτελούσε επικαιροποίηση των οδηγιών 10 χρόνια μετά, είναι ευκαιρία αυτή, για στήριξη περισσότερων δικαιωμάτων, παγίωση νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα υπήρχε και μια δυνατότητα συζητισμού της οδηγίας αυτής με άλλες σχετικές οδηγίες και με σαφήνεια στον τομέα παραδείγματος χάρη γονικής αδείας, μερικής απασχολήσεως, οδηγίας για εγκυμοσύνη και για συμβάσει ορισμένου χρόνου. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα πολύ συχνά και συμβιβασμοί που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να υιοθετηθεί και να εγκριθεί η νομοθεσία. Οι τροπολογίες θα πρέπει να συνάδουν με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όμως αυτή η ομολογία πολύ συχνά είναι τυχαία και δεν είναι συνεπής, είναι κατά περίπτωση. Και οι υποχρεώσεις των κρατών, κρατών μελών θα πρέπει να αναφέρονται σαφέστατα, κατά την άποψή μου. Επιπλέον, καμιά φορά πρέπει να ασχοληθούμε με οδηγίες που εφαρμόζουν συμφωνίες πλαίσια των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων. Και αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί που μπορούν να τροποποιούν αυτές τις συμφωνίες πλαίσιο, όπως η οδηγία για τη γονική άδεια. Αν έχετε σε στόχο νέα νομοθετική πρόταση, θα είχα τις εξής συστάσεις να σας κάνω. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τις υποχρεώσεις περιεφαρμογής που υπέχουν τα κράτη-μέλη, κάτι που δεν ήταν σαφές στην προηγούμενη οδηγία. Να συμπεριφθούν αναφορές σε διεθνές δίκαιο. Να γίνουν αποδεκτές πολλαπλές διακρίσεις και διατομεακές τέτοιες. Να υπάρχει διάταξη για την ταυτότητα των φίλων σε, σε συγκεκριμένες θέσεις που αφορεί, αφορά διάκριση σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου. Απαιτούνται δι, ε, ε, διευκρινήσεις για την εφαρμογή της αρχής της σύσης αμοιβή, κωδικοποιώντας την ομολογία, ανέφερα κάποια θέματα, Φερρυπίν. Η διάκριση στον τομέα αμοιβών ανδρών γυναικών απαγορεύεται, ανεξάρτητα από το σύστημα που οδηγήσετε τις διακρίσεις. Είτε είναι νομοθεσία, εφαρμογή ε, συνταξιδοτικών, τα συνταξιδοτικά συστήματα, εφαρμογή ε, των διαφόρων οδηγιών, εφαρμογή της αρχής οδηγίας. Δηλαδή η αρχή της ίσα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε στοιχείο της αμοιβή ξεχωριστά. Να τονίσω ότι η διαφάνεια περί αμοιβών θα πρέπει να τονιστεί όλος ιδιαίτερος, θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί, να κωδικοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις, τροποποιώντας τες ενδεχομένως οι διατάξεις των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Μαρτίου του 2014 περί διαφανείας αμοιβών. Θα μπορούσατε να εξετάσετε και τον δεχόμενο, να εξετάσετε πώς οι διαδικασίες ε, υπεργολαβιών και αναθέσεων μπορούν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογή της ε, οδηγίας. Θα τόνιζε επίσης και την ανάγκη που υπάρχει για μια συνεπή, συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τους διάφορους παράγοντες ε, με βάση το φύλλο και ε, την οδηγία για την κοινωνική ασφάλιση σύμφωνα με την ομολογία των δικαστηρίων. Συνταξιδοτικά συστήματα είναι αρκετά διαφορετικά στις διάφορες χώρες. Δεν γνωρίζουμε όλες οι χώρες το σύστημα των τριών πυλών που γνωρίζουμε εμείς. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Νομίζω επίσης ότι και οι διατάξεις περί αδειών θα μπορούσαν να εξεταστούν ξεχωριστά και να αναφερθούν ξεχωριστά και να υπάρχει ένα νέο νομικό μέσο σχετικά ίσως. Χρονικά όρια. Η νομολογία του δικαστηρίου δεν έχει κωδικοποιηθεί όσον αφορά το θέμα αυτό και δικαιώματα ενημέρωσης εκείνων που ζητούν εργασία είναι κάτι σημαντικό κατά τη δική μου άποψη. Αν επιλέξετε τελικά να μην κινηθείτε προς νέα πρόταση για νέα οδηγία, Υπάρχουν βέβαια και τρόποι και μέσα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της οδηγίας. Ανέφερα κάποιες λύσεις να ενισχυθεί η συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στην ομοθεσία και να παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη-μέλη σχετικά με αυτό. Αυτό θα ήταν σημαντικότατο. Φερρυπίν, αναπτύσσοντας και διαδίδοντας περαιτέρω αξιολογήσεις συνεπειών με βάση την ισότητα των φύλων και ε, διάφορα εργαλεία για τη χρηματοδότηση αυτών. Να πρέπει να τονιστεί περισσότερο η πρόληψη της ε, διάκρισης και αυτό συνεπάγεται και την καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Αυτό μπορεί να γίνει υπό το φως του άρθρου 5 της Συμβάσεως για την εξάλληψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, Φερρυπίν, που αναφέρεται στα στερεότυπα με βάση το φύλλο θα μπορούσατε να τονίσετε ότι τα αποτελέσματα που επιδιώκονται από την οδηγία είναι η ουσιαστική ισότητα. Αυτό αφορά και την ομολογία του δικαστηρίου άλλωστε. Και θα μπορούσατε επίσης να διαδώσετε και πληροφορίες περί απαγορεύσεως αλλαγής θέσεων με βάση το φύλλο. Δηλαδή ότι διακρίσεις με βάση την εγκυμοσύνη απαγορεύονται. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαγόρευση και οι οικονομικές συνέπειες της διάκρισης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξηγήσει και δικαιολογήσεις για την διάκριση. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες πληροφορίες για την ε, διαφάνεια των αμοιβών ε, όπως κωδικοποιείται από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προανέφερα Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να εντοπίσετε περαιτέρω κενά που υπάρχουν όσον αφορά την ε, προστασία των αυταποσχολούμενων γυναικών, όλους ιδιαίτερους, διότι διάφορες οδηγίες δεν παρέχουν επαρκή προστασία. Θα μπορούσατε να τονίσετε και τον ρόλο των φορέων ισότητας, κυρίως την ανεξαρτησία αυτών και ότι θα πρέπει να έχουν αρκετούς πόρους για την εκπλήρωση των σκοπών τους. Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν ε, βραχυπρόθεσμα. Να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες τελικά περί της ενδελεχούς έρευνας που διεξήχθη σε έξι Γαλλία, Λετωνία, Σλοβακία, Σπανία, Ολλανδία και Σουηδία ήταν οι χώρες. Και η επιλογή αυτών των χωρών βασίστηκε στο μέγεθος των χωρών. Θέλαμε παλιά και νέα κράτη-μέλη και θέλαμε επίσης και γεωγραφική ποικιλομορφία. Οι περιλήψεις των ερευνών αξίζουν τον κόπο να διαβαστούν, συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση, διότι μας έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίες αυτά τα προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη, κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση αυτής, σκοπός πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ορισμούς, έννοιες όπως άμεση και έμεση διάκριση και τα διάφορα προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή των ενιών, την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας και εν τέλει η έκθεση περιέχει συγκεκριμένες συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους εμπλεκομένους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους εθνικούς νομοθέτες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι Διεθνείς ε, έρευνες δείχνουν την ποικιλομορφία που υπάρχει όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κράτη-μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Το νομικό πλαίσιο ποικίλει από χώρα σε χώρα, στη Γαλλία, Φερρυπίν και στην Ισπανία όμως η οδηγία εφαρμόστηκε μέσω νέου νομοθετήματος και διατάξεις σχετικά με την ίση αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση θα βρεθούν σε πολλές πηγές. Αντιθέτως στην Ολλανδία δεν υπάρχει ανάγκη για θεωρήθηκε δεν χρειάζεται περαιτέρω, ε, να λυθούν περαιτέρω μέτρα για την εφαρμογή. Οπότε η εφαρμογή ε, της οδηγίας στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολλοί εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι υπήρχαν προβλήματα που σχετιζόταν με την απόδειξη της ε, διάκρισης. Ελπίζω ότι αυτό το έγγραφο παρέχει χρήσιμες συστάσεις, όλος ιδιαιτέρως για την εισηγήτρια επ' αυτού του θέματος και ανάλογα με το τι θα αποφασίσετε, ε, αν θα αναπτύξετε νέες προτάσεις ή θα προτείνετε περαιτέρω μέτρα για την επιβολή της οδηγίας από όλους τους φορείς, ε, ελπίζω να σας βοηθήσει αυτό το έγγραφο. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε στην δεύτερη ομιλητρία Ματζελεκούση, από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης που αναλύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων για το χάσμα το μισθολογικό Κύριε Δόκτωρα Κούρση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστώ τους διερμηνείς. Πολύ συχνά σε άλλα βήματα αισθανόμαστε την απουσία των διερμηνέων. Λοιπόν, εγώ τι θέλω να καλύψω. Θέλω να σας δώσω κάποιες ενδείξεις όσον αφορά την ε, έννοια της αμοιβή, πώς καλύπτω την οδηγία και να κινηθώ σε δύο κατευθύνσεις. Επιτρέψτε μου να πω παραδοσιακή κατεύθυνση καταρχάς των διαφορών όσον αφορά τις αμοιβέ. Πολλές φορές συζητούνται εδώ, πολύ συχνά συζητείται και στην οικονομική, στα οικονομικά κείμενα, συζητείται πολύ συχνά και σε πλαίσια εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ε, στους φορείς τους διεθνείς. Και θέλω να συνοδεύσω λοιπόν αυτό το θέμα με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των συντάξεων ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη, διότι οι συντάξεις, ε, σύμφωνα με την οδηγία, οδηγία δεν θα το επαναλάβω, μιλώ πάντα για την οδηγία 54 του 2006, ξεκινώντας από την έννοια της ε, αμοιβή. Λοιπόν, από αυτή την έποψη, λοιπόν, έχω συγκεκριμένες προτάσεις και παρουσίαση να κάνω, που αφορά καταρχήν κάποια στοιχεία που πρέπει να προσέξετε. Κάποια στοιχεία που θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και να δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο. Ελπίζω να είναι χρήσιμα τα στοιχεία λοιπόν που θα σας δώσω. Το πρώτο πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η ανάγκη που υπάρχει για στοιχεία που να είναι εύκολα προσβάσιμα και να είναι ομοιογενή, ούτως ώστε να γίνεται σύγκριση μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τα θέματα αυτά. Από την άποψη της αναλύσεως που έκανα, εγώ είδα ότι έπρεπε να εξετάσω δύο μεγάλες βάσεις δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χάρη στη δουλειά που έκανε το Ευρωστάτ. Είναι η βάση δεδομένων παραδοσιακά που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των δικτών της διαφοράς των πληρωμών ανάλογα με το φύλλο, δηλαδή διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τις αμοιβέ μεταξύ των δύο φύλων και το Stock Survey, δηλαδή τα στοιχεία που αφορούν τις αμοιβέ που γίνεται σε κάθε κράτος μέλος υπό το συντονισμό της Eurostat. Όμως πέρα από αυτή τη βάση δεδομένων που χρησιμοποιούμε ευρέω στα πλαίσια της ε, οικονομίας είναι και το ίκρα που δείχνει τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τα εισοδήματα και όσον αφορά τους ε, συνθήκες διαβίωσης ε, των Ευρωπαίων πολιτών διότι χάρη στην χρήση αυτού, του, αυτής της δεύτερης βάσης δεδομένων καταφέρουμε να έχουμε δείκτες πιο καλά στοχευμένους για να καταλάβουμε ε, τι οδηγεί στις διαφορές και τι συνέπειες έχουν οι διαφορές των αμοιβών και καταφέρνουμε πάνω απ' όλα να εντοπίσουμε τις διαφορές με βάση το φύλλο όσον αφορά τις συντάξεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δείκτης που να έχει δημιουργηθεί από το Ευρωστάτ όσον αφορά τις διαφορές ε, των, ε, των αμοιβών των φύλων στα πλαίσια της σύνταξης. Για την άποψή μου είναι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να προσεχθεί και να τονιστεί όταν επαναξεταστεί η οδηγία, διότι χωρίς τα στοιχεία προφανώς είναι δύστιχο να γίνει οποιαδήποτε εργασία ελέγχου και παρακολούθησης. Λοιπόν, σας δώσω μια ιδέα τώρα που οδηγεί αυτή η διαφορά μεταξύ των βάσεων δεδομένων και γιατί είναι σημαντικό να επιμένουμε επιχρήσεως στοιχείων που ταιριάζουν με την οδηγία από την άποψη του ελέγχου της εφαρμογής οδηγίας. Βλέπετε στο γράφημα ε, που προφανώς θα το βρείτε και στην έκθεσή μας και βλέπετε τις διαφορές αριθμητικές μεταξύ του δίκτυ διαφοράς των φύλων όσον να τις αμοιβές, να επενθυμίσω, είναι το gender pay gap αυτό, δείχνει το γράφημα, GPG έχει το γράφημα, που χρησιμοποιείται στις άλλες εκθέσεις, από το Gender Pay Gap, χρησιμοποιείται και από την ε, Διεύθυνση Έρευνας του Κοινοβουλίου. Βλέπετε διάφορα επίπεδα GPG διαφορών με βάση το φύλλο. Έχουμε με βάση δεδομένων το SILK και το SES, ε, το SES. E και βλέπετε διαφορά. Βλέπετε ότι τα επίπεδα είναι διαφορετικά με τις διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Τα στοιχεία SILK βλέπουν τη διαφορά των αμοιβών με βάση το φύλλο από το, που φτάνει το 31,1% ε, σε σχέση με το 16,4% των στοιχείων που ε, βρίσκονται και σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Κοιτάξτε και τη δυναμική με βάση το χρόνο. Εγώ στην ανάληψή μου κάλυψα την περίοδο μετά την εφαρμογή της οδηγίας, δηλαδή από το 2006 μέχρι το 2012 Δυστυχώς δεν έχουμε πιο πρόσφατα στοιχεία από το 2012 και πέρα. Ε, βλέπετε στην πραγματικότητα οι παραδοσιακοί δείκτες που βρίσκεται και στο σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ουσιαστικά την πορεία σχετικά σταθερή από 17,7 το 2006 και φτάνουμε στα 16,4 το 2012, ενώ στην πραγματικότητα τα στοιχεία SILK ε, σε υψηλότερα επίπεδα δείχνουν μειωτική τάση από 35 στο 31,1 πιο σημαντική διαφορά και πιο σημαντικά τα ποσοστά. Βλέπετε το πράσινο τετράγωνο που δείχνει τη διαφορά των φύλων όσον αφορά ε, τη σύνταξη. Έχουμε 38,3%, 38,3% επίπεδα, έχουμε και πιο υψηλά επίπεδα, 38,6% το 2010. Επίπεδο ουσιαστικά σταθερό τα τελευταία χρόνια, σχετικά σταθεροποιημένο, ε, χωρίς βελτίωση όσον αφορά τα στοιχεία ε, και αυτό είναι σημαντική αφετηρία για το προβληματισμό που θα ακολουθήσει. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κατά την άποψή μου το Gender Pay Gap, δηλαδή το GPG και το Gender Pension Gap, δηλαδή το GPG ε, και τα δύο στοιχεία είναι συνιστός βασικές της έννοιες των αμοιβών. Σε όλη μου την ανάλυση έλαβα υπόψη και τις δύο συνιστώσεις από ό,τι γνωρίζω ποτέ δεν έχει γίνει πριν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ε, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία που αναπτύξαμε με βάση τη βάση δεδομένων SILK. Δεν έχω το χρόνο να σας δείξω όλα τα αποτελέσματα. Ελπίζω ότι θα έχετε τη βούληση και την χαρά να διαβάσετε την έκθεσή μας. Εν πάση περιπτώσει, τα αποτελέσματα από την ε, οπτική γωνία των χαρακτηριστικών των διαφόρων που προσμετρήσαμε είναι εξαιρετικά σημαντικά και ενδιαφέροντα. Το gender pay gap είναι πολύ πιο μεγάλο για τους ε, μερικά απασχολούμενους από ότι τις εργαζόμενους πλήρης απασχόλησης. Το ίδιο αφορά και τη διαφορά με βάση τις συμβάσεις, κυρίως οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου. Ε, ε, εκεί υπάρχει διάκριση όσον αφορά την αμοιβή. Το gender pay gap οι διαφορέ με βάση το φύλλο όσον αφορά τι αμοιβέ αυξάνονται με την ηλικία. Αν αναλύσετε τον κύκλο ζωή, επιδεινώνονται με την ηλικία των ατόμων και δεν βελτιώνονται. Ξεκινάνε πιο κοντά τα, οι αμοιβέ και μετά απομακρύνονται και η ηλικία αφορά και σωρευμένε γνώσει όσον αφορά και εμπειρία από την εργασία. Και άρα θα υπήρχαν και πολλά κινήτρα αυξημένα για την αύξηση τη πληρωμή και υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορέ όσον αφορά τα τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης και του τομείς απασχόλησης. Αυτό προφανώς μας οδηγεί να ε, σταυρώσουμε το θέμα της, του διαχωρισμού ε, και της απομόνωσης που θα αναλύσω αργότερα. Πριν περάσω τώρα στο gender gap στις συντάξεις, δηλαδή τις διαφορές όσον αφορά τις συντάξεις με βάση το φύλλο, σας δείξω ένα άλλο γράφημα ε, που αφορά τις διαφορές των αμοιβών. είναι ένα αποτέλεσμα που ήδη έχουμε βρει, να σας το δείξω με χαρά. Λοιπόν, ξανά η περίοδος 2006-2012, ε, ο δημόσιο τομέα, κάνει τη διαφορά λοιπόν εδώ. το εργάζεται κανεί στο δημόσιο τομέα, δεν εξαλείφει τις διαφορές. Στον τομέα το δημόσιο ε, υπάρχουν πολύ περισσότερα κίνητρα να υπάρχει διαφορά, αλλά μειώνεται. Υπάρχει μια προστασία λοιπόν όσον αφορά τη δουλειά των γυναικών στις θέσεις που υπάρχουν εντός του δημόσιου τομέα και αυτό οδηγεί σε μείωση της διαφοράς ή εξάγονται στον ιδιωτικό τομέα, ίσως θα εξαχθούν στον ιδιωτικό τομέα εγγυήσεις που παρέχονται στο δημόσιο τομέα. Αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί μέσω ισχυρής συμμαχίας μεταξύ συνδικάτων ή όλων εκείνων που εργάζονται στον τομέα των βιομηχανικών σχέσεων, των σχέσεων στον τομέα της εργασίας. Λοιπόν, στις συντάξεις έχουμε το gender gap, ε, είδαμε ότι είναι πολύ μεγάλε οι διαφορέ, πολύ μεγαλύτερε σε σχέση όσον αφορά τι αμοιβέ των εργαζομένων. Άλλη διάκριση που θα ήθελα να σα δείξω αφορά την φύση των συντάξεων, διότι γνωρίζουμε καλά ότι τα τελευταία χρόνια πολλέ μεταρρυθμίσει του ταξιδιωτικού τομέα έχουν επηρεάσει ε, μέσω της αγωγής δεύτερου πυλώνα σε κάποιες χώρες, υποχρεωτικά έχει εισαχθεί δεύτερος πυλώνας όσον αφορά τις ιδιωτικές συνταξιδοτήσεις. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία που σας δείχνω τώρα, παρακαλώ να δείτε πώς υπάρχουν διαφορές με βάση το φύλλο όσον αφορά τις συντάξεις που έχουν τονιστεί, έχουν αυξηθεί όταν επικεντρωθεί κανείς στις συντάξεις του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τις δημόσιες συντάξεις. Ε, βλέπετε λοιπόν τρία γραφήματα, τρεις γραμμές και οι τρεις γραμμές αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς δεν έχω το χώρο και το περιθώριο να σας δείξω όλα τα, τα αποτελέσματα κατά χώραν. Μπορώ αν το ζητήσετε. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία στα γαλάζια που είναι τα στοιχεία που σας έδειξα που είναι από το 38,3 το 2012 και βλέπετε και τα προηγούμενα στοιχεία. Μετά βλέπετε στα πράσινα μια γραμμή που αφορά εκείνους που έχουν μόνο ιδιωτική συνταξιδότηση και όχι δημόσια και ιδιωτική, μόνο ιδιωτική σύνταξη και ήδη αυτό μας οδηγεί πολύ πιο ψηλά, δηλαδή το 2011 μας σε επίπεδο διαφοράς που φτάνει το 52,3% και μετά αν δείτε εκείνους που έχουν συντάξεις και δημόσιες και ιδιωτικοί αλλά επικεντρωθούμε επί της συνιστώσας της ιδιωτικής αυτού του ε, μεικτού εισοδήματος οι διαφορές είναι συντριπτικές τεράστιες. Έχουμε διαφορές του ύψους του 70%. Είναι άχρηστο να υπογραμμίσω τι οδηγεί σε αυτό το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο έλλειψης δυνατότητας από των γυναικών να συνεισφέρουν συνεχώς στα συνταξιωτικά ταμεία του ιδιωτικού τομέα και θα αναφερθώ σε αυτό και σε μια κοινή ανάλυση των δύο δικτών. Ε, τώρα εντάχει φτάνω λοιπόν στην ολοκλήρωση. Έκανα μια μελέτη μεικτή των δύο δικτών για να μπορέσω να δείξω ποια μπορεί να είναι τα στοιχεία τα κοινά ε, που οδηγούν στα προβλήματα τα οποία διαπιστώσαμε. Ένα πράγμα θέλω να σας ε, δείσω στις διάφορες μεταβλητές που εξέτασα στην οικονομητρική ανάλυση έβαλα και μια μεταβλητή που δείχνει και τι γίνεται όσον αφορά την πρόσληψη της οδηγίας, πώς εφαρμόστηκε η οδηγία σε διάφορες χώρες. Λοιπόν, ε, έλαβα υπόψη και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013 όσον αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής μέχρι τότε. Λοιπόν, ε, βλέποντας λοιπόν αυτή την τεκμηρίωση που έλαβα υπόψη και βλέποντας τις χώρες που έχουν ενσωματώσει και έχουν υλοποιήσει την οδηγία με αυτή τη μορφή σε όλες τις χώρες που έχουν εφαρμόσει την οδηγία σύμφωνα με την έκθεση αυτή βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση και του gap όσον αφορά τις αμοιβέ και του gap όσον αφορά τις συντάξεις. Λοιπόν, μετά βέβαια αυτά τα αποτελέσματα βάλαμε και άλλες θεσμικές μεταβλητές ε, στην έρευνα που κάναμε και στην ανάλυση που κάναμε που λαμβάναμε υπόψη τις διαφορές που υπήρχαν όσον αφορά την εκπαίδευση, τη δομή της απασχόλησης, της ηγετική θέση που έχουν οι γυναίκες στον τομέα, πώς ώρες εργάστηκαν και την παρουσία των μεταναστών και διάφορες μεταβλητές ταξινόμησης, ranking, που λάβαμε υπόψη από το Ευρωπαϊκό ε, Institute to Gender Equality και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμποποιηθούν στην ανάλυση αυτού του τύπου που πρέπει να γίνεται και σε άλλα πλαίσια το European Institute of Gender Equality έκανε πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά τη δημιουργία νέων δικτών ε, και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες αυτούς ε, και αναλύσαμε και τον ρόλο των minimum wages όπως θα δείτε σε λίγο είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Είναι σημαντικά τα minimal wages όσον αφορά την μείωση της, ε, του gender gap στις συντάξεις οπότε παρέχεται μια προστασία της νομοθεσίας και των διατάξεων όσον αφορά τα ελάχιστα εισοδήματα ε, των εργαζομένων και αν γίνει αυτό θα ήταν ε, μια κίνηση προς την ευκταία κίνηση, δηλαδή να μειωθούν οι διαφορές. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να σας δείξω όλα τα αποτελέσματα, όμως ε, προφανώς κατόπιν ετήματος μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Τι είδους συστάσεις μπορούν να βγουν από την έκθεσή μου σχετικά με την δουλειά που κάνετε εσείς οι τομείς παρέμβασης είναι οι ίδιοι που αναφέρονται επανειλημμένως. Πρώτα απ' όλα η έκθεση Bauer που ελήφθηκε σαν σημείο αναφοράς ε, για τις παρατηρήσεις μας είναι η βάση. Δεν θα αναφέρω τα ίδια που αναφέρεται στην έκθεση αυτή, αλλά πολύ πιο συγκεκριμένα πιστεύω ότι είναι υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να στερνιστεί όλες τις αποκομιστήσεις εμπειρίες στον τομέα αυτό, τους πειραματισμούς, να συλλέξει, να συνεθρήσει τις εμπειρίες του παρελθόντος και του παρόντος πιστεύω ότι είναι ένα λάτωμα που πολύ συχνά ε, μας διακρίνει στην ανάλυση να ξεκινάμε πάντα από την αρχή σαν να μην έχει γίνει τίποτα εκ του μηδενός. Όμως είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε όλα αυτά που έχουν γίνει, ό,τι έχει οριμάσει σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό, τομεακό και οργανωτικό. Και πιο, πιο συγκεκριμένη σκοπιά των διαφόρων λεπτομεριών της παρέμβασης είναι σημαντικό και κάτι που γραμμίστηκε από την προλαλή σας συνάδελφο να εντοπίσουμε τους συγκεκριμένους targets, στόχους. Θα ήθελα χάρη στις δικές σας παρεμβάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να καθορίσει targets προς επίτευξη από μια οπτική γωνία χρονική και όσον αφορά το gender pay gap και το gender pension gap. Να αυξηθεί η διαφάνεια να εισαχθούν διάφορες μορφές καταπολέμησης της ε, διάκρισης και σίγουρα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε αργότερα. Ποιος είναι ο δικός σας ρόλος ε, να αυξηθεί η επίγνωση όσον αφορά του θέματος και ευαισθητοποίηση και να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σε μια έκθεση σε άμεση επαφή με τα κράτη-μέλη να καταρτήσει κάποια μέθοδο ανοιχτού συντονισμού, όπως ήδη έγινε και για τις ε, συντάξεις, αλλά με συγκεκριμένο τρόπο όσον αφορά τη διαφορά των φύλων. Κλείνω υπενθυμίζοντας ότι το 2012 το Pension Adequacy Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη υπογράμμισε το πώς η βασική πρόκληση και στόχος για τις συντάξεις στο μέλλον, το εγγύς μέλλον, είναι να μπει η πτυχή των φύλων. Η νέα έκθεση που Μάιο-Ιούνιο θα βγει νομίζω ε, η Pension Adequacy, Report θα με ενδιαφέρει να δω πώς θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Θέλω να το δω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόρση. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το κατάλογο των ομιλητών πρωτού ακούσουμε τις ερωταπαντήσεις. Άρα να ακούσουμε και τους τέσσερις ομιλητές και μετά να περάσουμε στις ερωταπαντήσεις. Η Τάνια λέει έχει το λόγο. Από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο που Βέλπε της δόκτωρα Βέλπε στην ομάδα της για την αξιολόγηση και κατάταξη των θέσεων απασχόληση. Um, ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα σε σχέση με την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας. Καταρχάς, τι περιλαμβάνει ο ορισμός των συστημάτων εξαλληλόγησης και κατάταξης των ε, θέσεων εργασίας ουδέτερων ω προ το φύλλο. θα δούμε πώ εφαρμόζονται αυτά τα κράτη-μέλη και θα κάνουμε κάποιε συστάσει για τη βελτίωση τη εφαρμογή. Στην οδηγία, η αρχή τη ε, εργασία τη αξία ορίζεται και ουσιαστικά αναφέρεται ότι τα, τα άτομα που εκτελούν ίδια εργασία ή στι αξίε εργασία θα πρέπει να λαμβάνουν τον ίδιο μισθό. Δηλαδή, ένας μηχανικός και μία γραμματέας που κάνουν ένα έργο ίσης αξίας θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον ίδιο μισθό. Πώς εκτιμούμε, πώς αξιολογούμε όμως το κατά πόσον η εργασία είναι ίσης αξίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης της εργασίας. Και τα συστήματα αυτά κυρίως κοιτάνε τις απαραίτητες προδιαγραφές, τις απαραίτητες απαιτήσει για μια θέση εργασίας. Οι ικανότητες, οι ευθύνε και ύστερα ε, καθορίζουν τα επίπεδα μισθού. Η οδηγία καθορίζει ότι αν χρειάζονται και αν χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα θα πρέπει να είναι ουδέτερα ως προς τη διάσταση του φύλου. Είναι ατυχές ότι λίγες είναι οι συστάσεις μέσα στην ίδια οδηγία για το πώς θα καταστούν ουδέτερα προς το φύλλο αυτά τα συστήματα. Αναφέρονται μόνο οι ίδιοι παράγοντες, οι ίδιες, τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να ισχύουν για γυναίκες και άντρες, ότι αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τα συστήματα αξιολόγησης εργασίας, ε, ουδέτερα προς το φύλλο, στο έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Μία πρώτη σύσταση όμως θα ήταν να συμπεριληφθούν αυτές οι συστάσεις σε ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας, προκειμένου τα κράτη-μέλη να έχουν ένα εργαλείο για την διαμόρφωση των συστημάτων με ουδέτερο προς τα φύλλα τρόπο. Σε ποιο βαθμό όλο τώρα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ήδη αυτό το σύστημα αξιολόγηση τη εργασία, Έξι χώρε. Γερμανία, Μάλτα, Σουηδία, Λεπτονία, Ηνωμένο Βασίλειο και το επίπεδο υλοποίησης είναι αρκετά χαμηλό. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν ήδη εκταμένες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς τα συστήματα θα είναι ουδέτερα προς το φύλλο. Σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς εταίρους, βλέπουμε ότι τα συνδικάτα είναι πιο ενεργά και δραστηρία παρά οι εκπρόσωποι των ε, εργοδοτών και υπάρχουν πιο πολλές ε, δραστηριότητες στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά τα σώματα ισότητας, βλέπουμε και εδώ μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Στη Λατωνία και στη Μάλτα δεν έχουμε εκτεταμένες δραστηριότητε, αλλά στην Γαλλία, Σουηδία και στον Εμένο Βασίλειο είναι ανεπτυγμένο το σκέλος αυτό. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει περιθεωρείο περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και κατάταξης θέσεων απασχόλησης και θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες συστάσεις για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Καταρχάς, θα συστήναμε να βελτιωθεί η οδηγία να συμπεριληφθούν πιο πολλές συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς τα συστήματα αυτά θα πρέπει να καταστούν ουδέτερα προς τη διάσταση του φύλου. Από επιστημονικής άποψης πολλά μπορούμε να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό. Για παράδειγμα, οι επιτροπές αξιολόγησης που αξιολογούν και εκτιμούν τις θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να είναι και αυτές ουδέτερες ως προς το φύλλο ή σε αντιπροσώπευση γυναικών και ανδρών με ε, εκπαίδευση σε ό,τι αφορά τα στερεότυπα, σε ό,τι αφορά το φύλλο. Γιατί αυτό συχνά οδηγεί σε υποτίμηση της δουλειάς των γυναικών και χαμηλότερο μισθό. Επίσης θα πρέπει να είναι υπεύθυνες αυτές οι επιτροπές για να δικαιολογήσουν και να τεκμηριώσουν τις αποφάσεις τους σε ενδεχόμενη περίπτωση ελέγχου. Αν συσταθεί λοιπόν μια τέτοια επιτροπή και υπάρχει περιγραφή θέσεων για κάθε θέση σε κάθε εταιρεία, θα πρέπει να αποφασίσουμε, θα αποφασιστεί ουδετερότητα και στην διατύπωση για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη χρήση γυναικείων ή άνδρικων ε, όρων στη γλώσσα. Και επίσης να ληφθούν υπόψη ε, οι διαστάσεις ε, των προσωπικών ενδεχομένω προβλημάτων. Κάποια στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να εκτιμηθούν, γιατί ο καθένας κατανοεί με διαφορετικό τρόπο ενδεχομένως διάφορες περιστάσεις και αυτό οδηγεί στην διαιώνιση των στερεοτύπων. Αν αυτοί οι παράγοντες λοιπόν οριστούν, μετά θα πρέπει να συλλεχθούν τυποποιημένα δεδομένα, τυποποιημένες συντεύξεις να δίδονται στους εργοδότες για να καθορίζεται σε ποιο βαθμό αυτοί οι παράγοντες, αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για μια θέση. Και αν υπάρχει λοιπόν, όταν διαμορφωθεί λοιπόν η περιγραφή της ε, κάθε θέσης, θα πρέπει να υπάρξει κάποια στάθμιση των ε, στοιχείων αυτών. Πόσο σημαντικό είναι, για παράδειγμα, το στοιχείο της ε, ευαισθησίας στα διαπροσωπικά προβλήματα σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι διαρκώς υποτιμούνται οι γυναικείες ικανότητες, όπως για παράδειγμα η ικανότητα επίλυσης διαπροσωπικών προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Επίσης, ο χαρακτηρισμός ε, θηλυκών και αρσενικών ικανοτήτων. Σε ένα τελευταίο βήμα, θα πρέπει να υπάρχει κατάταξη της θέσης ανάλογα με τη μισθολογική της αξία. Αυτό είναι σημαντικό να γίνεται προτού ξεκινήσει η εργασία. Από πριν λοιπόν θα πρέπει να αποφασίζεται σε τι βαθμούς θα πρέπει να φτάσει μία θέση εργασίας σε ένα μισθολογικό επίπεδο. Γιατί γενικά υπάρχει τάση οι γυναίκες να κατατάσσονται σε χαμηλότερο μισθολογικό επίπεδο. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, θα υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης ε, της θέσης και αυτό θα βελτιώσει το μισθολογικό χάσμα. Ωστόσο, οι περιγραφές των θέσεων απασχόλησης που ε, δημιουργήθηκαν μέσω αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να, την, να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε κάποιες θέσεις απασχόλησης με, την, τον ορισμό αυτών των παραγόντων και υποπαραγόντων για τη διαδικασία επιλογής, για την εκτίμηση των ικανοτήτων κάποιου υποψηφίου και το καθεξής. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες στο σημείο αυτό, αλλά αν σας ενδιαφέρει περαιτέρω συστάσεις μπορείτε να τις βρείτε στην έκθεση της μελέτης μας. Επιπλέον, θα θέλαμε να συμπληρωθεί η οδηγία σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το μισθό. Τα συστήματα αξιολόγησης εργασίας υποθέτουν ότι δεν γίνεται καθορισμός του μισθού βάσει της απόδοσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα άλλαζαν τα συστήματα και ξέρουμε ότι στις διαπραγματεύσεις ε, για το μισθό όταν ε, οι γυναίκες ζητούν αύξηση πολλές φορές αυτό ε, γυρνάει μπούμεραγκ και για παράδειγμα δεν παίρνουν τη θέση αυτή. Η απόδοση των γυναικών συχνά αξιολογείται χαμηλότερη σε σχέση με τον ανδρών λόγω στερεοτύπων αναφορικά με το φύλλο. Γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να είναι ουδέτερες και διαπραγματεύσεις ανάλογα με το φύλλο και να υπάρχει μισθός ανάλογα με την απόδοση. Περισσότερες λεπτομέρειες και πάλι μπορείτε να βρείτε στη μελέτη μας. Θα σας στείναμε επίσης προώθηση, περαιτέρω προώθηση την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στα κράτη-μέλη. Και στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη και η κοινωνική τους εταίροι και τα σώματα ισότητας να αναπτύξουν εργαλεία αποτροπής προκειμένου να αναπτυχθούν συστήματα με ισότητα ως προς την διάσταση του φύλου. Γιατί συχνά το πρόβλημα είναι ότι οι οργανώσεις δεν ξέρουν πώς να διαμορφώσουν συστήματα ουδέτερα. Άρα, κατευθυντήριες γραμμές, ε, κατάλογοι και επιπρόσθετα θα μπορούσαν να υπάρξουν εθνικοί εθνικές αλλά και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων όπου θα αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία και αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα χρειαζόταν κάθε μεμονωμένη εταιρεία να κάνει αξιολόγηση βάσει των συστημάτων αυτών. Εν συντομία τώρα για την τελευταία μας σύσταση για την παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας πιστεύουμε ότι θα ήταν σημαντικό αυτό ε, να γίνει μια μελέτη στα κράτη-μέλη που θα αξιολογεί συστηματικά σε ποιο βαθμό οι οργανώσεις ήδη εφαρμόζουν τα συστήματα αξιολόγησης ε, εργασίας και σε ποιο βαθμό είναι ουδέτερα τα συστήματα που εφαρμόζουν. Αυτό θα βοηθούσε για την ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας. Γιατί αυτό θα ε, επέτρεπε, θα να εξετάσουμε κατά πόσον είτε ήδη επιτυχημένη η οδηγία. Έτσι, ενδεχόμενη μεταρρύθμιση, αναθεώρηση της οδηγίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκριση των αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ και έρχεται και τα στοιχεία επικοινωνίας μου σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν. Η Πρόεδρος δίνει το λόγο. Στην κυρία Τσέλεβα από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας σε ό,τι αφορά τις άδειες μητρότητος και πατρότητος σε ό,τι αφορά θέματα ισότητας των φύλων. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Μία ερώτηση, μια και περιμένουμε. Θα μπορούσαμε να λάβουμε τις διαφάνειες, γιατί κάποιες από τις διαφάνειες δεν προλάβαμε να τις διαβάσουμε, δεν ήταν εύκολο να τις διαβάσουμε από εδώ. Η πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι. Θα παρακαλέσουμε τη Γραμματεία να μας τη διαβιβάσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ο ρόλο μου εδώ ήταν να κοιτάξουμε ε, την εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας, αλλά σε ό,τι αφορά την άδεια τη γονική, τη μητρότητος και εδώ κοιτάξαμε κυρίως τρεις διατάξεις, τις γενικές διατάξεις που ορίζουν την λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των γενικών σε σχέση με την εγκυμοσύνη, με την αδεία μητρότητος ως μορφή διακριτικής μεταχείρισης και δύο συγκεκριμένες λοιπές διατάξεις για την προστασία των ε, ατόμων που επανέρχονται στη θέση, ε, στη, στη εργασία τους μετά από κάποια τέτοια άδεια. Κυρίως την άδεια μητρότητος, άρθρα 15 ή 16, ε, την πατρική άδεια και την άδεια υιοθεσίας. Κοίταξα και την μεταφορά της οδηγίας στα εθνικά νομικά συστήματα, αλλά αυτό που με ενδιέφερε ακόμα πιο πολύ ήταν ο κοινωνικός αντίκτυπος των διατάξεων. Κυρίως σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των νομικών διατάξεων στα εθνικά νομικά συστήματα. Προσπάθησα να εντοπίσω τις διάφορες προκλήσεις. Το πρώτο τμήμα των προκλήσεων. Εξετάσαμε ζητήματα προστασίας και το εύρος της προστασίας. Κατά πόσον η προστασία είναι ρητή στα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Εδώ διαπιστώσαμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τον ορισμό της προστασίας, κατά πόσον καλύπτει όλους τους εργάτες και εργαζόμενους. Κατά πόσον ήταν πλήρη η μερική προστασία. Για κάποια κράτη-μέλη διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα. Ένα δεύτερο πρόβλημα τώρα ήταν στο θέμα της απόλυσης και της ε, δυνατότητας αγωγής μετά από απόλυση. Πρό, πρόσβαση λοιπόν στα ένομα 11 μέσα. Για άτομα τα οποία έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση, εδώ είχαμε προβλήματα σε ό,τι αφορά το βάρος απόδειξης, αλλά και σε ό,τι αφορά το υψηλό κόστος της αγωγής. Κάποιες από τις δικαστικές ε, ένομες ε, τέτοιες ε, διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και αυτό μειώνει μοιραία τον ρυθμό των ατόμων που ενδεχομένως να προσπαθήσουν να προβάλλουν αξιώσεις έναντι του εθνικού συστήματος καθώς και την πιθανότητα αποζημίωσης μετά από απόλυση ή διακριτική μεταχείριση. Αλλά θετικά στοιχεία πρέπει να σας πω ότι έχω εντοπίσει και κάποιες καλές πρακτικές, κάποιες χώρες όπου η προστασία των εργαζομένων είναι ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται από την οδηγία μετά από μητρική η γονική άδεια. Στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα τρίτο μέρος παρόν όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία απόλυσης ευάλωτων, ευαίσθητων εργαζομένων στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει, να είναι παρόν δημόσιος ε, υπάλληλο για να εγγυόμαστε την ισορροπία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα νομικά συστήματα λειτουργούν με προβλήματα, με ελαττώματα, υπάρχουν πολλά πιο πολλά προβλήματα, πολύ πιο πολλά προβλήματα στην εφαρμογή, στην υλοποίηση των διατάξεων. Υπάρχουν λοιπόν κενά μεταξύ της νομοθεσίας και της πράξης και εδώ δεν έχουμε δεδομένα. Είναι πολύ κατακριματισμένα και ελλειπή τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξέρουμε όμως ότι σε κάποιες χώρες 10% των γυναικών απολύονται μετά την αδιαμετρότητα. Έχουμε στοιχεία σχετικά από την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε Ιταλία, Τσεχική Δημοκρατία, Πορτογαλία, οι χώρες, οι γυναίκες δέχονται πίεση για να παρατηθούν, εθελούσια. Αυτό ονομάζεται λευκή απόλυση, παρέτηση. Είναι όμως ε, αρκετά ελλειπή τα στοιχεία αυτά. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να, να καταγραφούν πιο πολλά στοιχεία. Ένα δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω. Το θέμα ενός ε, μιας ε, μιανεκτούσας μερίδας των εργοδοτών. Φυσικά υπάρχουν νομοθεσίες που προστατεύουν τους εργαζόμενους και επίσης οι συμβάσεις ορισμένης διάρκειας συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα τον εργασιακό. Αλλά τι γίνεται με τις μητέρες, για παράδειγμα, που δεν ε, ανανεώνουν τα συμβόλαιά τους μετά την αδιαμητρότητα. Τι γίνεται με τις γυναίκες που απασχολούνται με κώδικα αστικού δικαίου. Αυτές εμπίπτουν ε, εκτός του πεδίου οποιαδήποτε προστασίας και οι Ευρωπαίοι πολίτες μας κάνει εντύπωση. Φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν ποια τα δικαιώματά τους. Περίπου 50% όλων των Ευρωπαίων πολιτών δεν γνωρίζουν, δεν αντιλαμβάνονται τα δικαιώματά του σε περίπτωση διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση. Λαμβάνοντα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη, Φυσικά έχω ένα μακρύ κατάλογο συστάσεων. Αυτό όμω που θα ήθελα τώρα να τονίσω είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλό θα ήταν να καλέσει τα κράτη-μέλη να παρακολουθήσουν τον αριθμό, τον χαρακτήρα των διακριτικών μεταχειρήσεων και την, ε, τη διαθεσιμότητα ένομων μέσων για την κατεπολέμηση τέτοιων περιπτώσεων διακριτική μεταχείριση. Επίση, ευαισθητοποίηση, προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτε να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν σε περίπτωση που του συμβεί κάτι τέτοιο. Ίσως και ότι υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω προστασίας ενός ε, μειονεκτούντος μεριδίου της ε, αγοράς εργασίας για τα μη, τυπικά, τυπικές συμβάσεις, για παράδειγμα, θα πρέπει να λεφθούν υπόψη οι συμβάσεις ορισμένης διάρκειας. Τέλος, η οδηγία για την ε, άδεια μητρότητας. Ίσως ε, να πρέπει να προσαρμοστεί και θα μιλήσω γι' αυτό και στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στο γύρο ερωταπαντήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε το δυνατόν πιο σύντομοι. Να ξεκινήσει ίσως η συγγήτρια. Κυρία Ζαμπόρφσκα, θέλετε να θέσετε κάποια ερώτηση, όχι? Δεν δεν έχω ακόμα ερώτηση. Η κυρία Μπίρντερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις εισηγήσεις σας. Είναι πραγματικά συναρπαστικές. Με ενδιαφέρον είδα πόσο αλλάζουν όλα αυτά τα στοιχεία από τη μία χώρα στην άλλη στην Ευρώπη. Η διαφάνεια των μισθών και το χάσμα που υπάρχει στις συντάξεις είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι μια ορολογιακή βόμβα. Όταν δεν έχουμε μισθολογική ισότητα τώρα, αυτό το πληρώνουμε πολύ αργότερα. Κανείς όμως δεν ανέφερε τις ε, διαδικασίες ε, παραπώνων, παραπτωμάτων, επιπαραβάση και το καθεξής. Στο Ηνωμένο ε, Βασίλειο έχει συμφωνηθεί ένας τέτοιος νόμος που αποτελεί μέρος η ρήτρα αυτή στην εκάστοτε σύμβαση. Και με ενδιαφέρον ανακάλυψα ότι αυτό δεν ισχύει στις άλλες χώρες. Όμως, σε, στο θέμα αυτό οι γυναίκες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι του ισχυρού άνδρα αφεντικού τους. Και πρέπει να βοηθηθούν στη διαπραγμάτευση αυτή. Κάτι άλλο που έχω σημειώσει είναι το εξή. Αναρωτιέμαι. Μήπως θα έχουμε τους δείκτες μετανάστευσης για να έχουμε καλύτερες διατάξεις για τις κρατικές συντάξεις αφού υπάρχει αυτό το χάσμα στις συντάξεις και ε, για τις γυναίκες που δεν θα μπορέσουν να κατακτήσουν το εξωτερικό δικαίωμα στη χώρα μέλος τους. Το έχετε σκεφτεί. Από εκεί και πέρα, η έλλειψη γνώσης, συνειδητοποίηση από πλευράς κοινο... κοινωνίας είναι τεράστιο πρόβλημα. Εγώ εργαζόμουν σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό, ε, ε, γραφείο παροχής συμβουλών σε πολίτες και ε, πραγματικά είδα ότι είναι απίστευτο το πόσο καθόλου δεν καταλαβαίνουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους και πόσο ευθύνη δικιά μας είναι να τους τα μάθουμε, ευθύνη των κυβερνήσεων. Πολύ συχνά δεν το κάνουν αυτό. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κυρία Μορφάη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ίση αμοιβή για ίση δουλειά. Αυτή η αρχή ήταν ήδη παρούσα στην ομοθεσία του 2006. Η ιστορία είναι μακρά. Εμφανίστηκε πρώτη φορά ο όρος στη δεκαετία του 70. Ε, είναι ένας υποχρεωτικός νόμιμος κανόνας, νομικός κανόνας. Η οδηγία είναι υποχρεωτική και πρέπει να την εσωματώσει το κάθε κράτος μέλος στην εγχώρια νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι όποια χώρα μέλος και αν εξετάσουμε είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου να μην υπάρξουν διαφορές στην πληρωμή, στην αμοιβή ανδρών και γυναικών. Ωστόσο, Ακούσαμε τώρα από τις εισηγήτριες ότι οι διαφορές παραμένουν και είναι σοκαριστικές στην αμοιβή ή πληρωμή ε, γυναικών ή ανδρών. Και το νιώθουν οι πολίτες, το βλέπουν με τέτοια τους τα μάτια, ότι στην ίδια δουλειά οι γυναίκες κερδίζουν πολύ λιγότερα από ότι οι άνδρες που κάνουν την ίδια δουλειά. Πώς είναι, εδώ, πώς είναι αυτό δυνατό. Είναι πολύ απλό το ερώτημα και θέλω να σας το θέσω. Πώς γίνεται αυτό. Δεν αντιφατικά αυτά τα δύο γεγονότα. Πώς γίνεται να είμαστε πάλι σε αυτή την κατάσταση. Από, την άλλη, από τη μία νόμος να μας υποχρεώνει ήδη από το 2006 για να μην μιλήσω για τη δεκαετία του 70 και τα κράτη-μέλη από την άλλη δεν τον τηρούν. Πώς γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατό. Θέλω απάντηση παρακαλώ. Και επίσης, άλλο ερώτημα. Τι γίνεται εάν κάποιος προσπαθήσει να ε, εξαναγκάσει έτσι ώστε να επιβληθεί αυτή η νομοθετική διάταξη. Ξέρετε, οι εργατικές διαφορές υπάρχουν και μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες εργαζόμενες δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για να στραφούν δικαστικά, να προσφύγουν στο δικαστήριο για να εφαρμοστεί ε, αυτή η νομοθετική διάταξη. Δίδεται στήριξη στις γυναίκες αυτές. Αυτές που υποφέρουν από διάκριση ούτως ή άλλως κερδίζουν πολύ λιγότερα και έχουν πολύ μικρότερα εισοδήματα. Υπάρχει στήριξη που δίδεται σε εκείνες τις γυναίκες για να μπορέσουν να κινηθούν δικαστικά, να ασκήσουν όλα τα ένδικα νόμιμα μέσα. Ποιες είναι οι ευκαιρίες που έχουν. Θα ήθελα να μπορώ να πω στις ψηφοφόρους μου, στην Ουγγαρία, πού μπορεί να πάνε, πού μπορούν να στραφούν, εάν δουν ότι ε, πληρώνονται λιγότερο για την ίδια δουλειά από ότι οι άνδρες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ε, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω σε ποια από τις εισηγήτριες, όμως η ερώτηση είναι η εξής. Οι διαφορές στην αμοιβή, στις θέσεις στην ιεραρχία και στις συντάξεις, όπου οι διαφορές είναι τεράστιες, εξόφθαλμες, οφείλονται μήπως στην έλλειψη τήρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή μήπως οφείλονται, και αυτό είναι άποψή μου, στο γεγονός ότι η περίοδος ανατροφής των παιδιών για τις γυναίκες δεν τη χάνει αντισταθμίσματος. Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε από το σύστημα που αναλύσατε, ότι δηλαδή οι γυναίκες ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα και αυτό τις κρατάει πίσω και τελικά αυτό είναι ε, ε, αυτό στο οποίο οφείλεται η μεγάλη διαφορά στις συντάξεις. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Κύρια Κόρση, μιλήσατε για την όξυνση των μισθολογικών ανισοτήτων στις θέσεις μερικής απασχόλησης και στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό το είδος εργασίας που είναι λιγότερο καλυμμένο, καλύπτεται λιγότερο αν θέλετε από τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και συλλογικέ συμβάσεις. Επίσης, οι επιθεωρήσεις, η επιθεώρηση εργασίας. Η κυρία Σέλεβα αναφέρθηκε στις απολύσεις εν λευκό για τις εγγύους ή τις εργαζόμενες μητέρες. Θα ήθελα να γνωρίζω, υπάρχουν επιθεωρητές εργασίας που επαληθεύουν ακριβώς τι συμβαίνει. Γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει, αλλά κανείς δεν πάει εκεί να εξετάσει. Άλλωστε οι μισθωτοί με χαμηλούς μισθούς που έχουν λιγότερη κατάρτιση γνωρίζουν λιγότερο και τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. σε ό,τι αφορά το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου για την έκθεση αυτή. Ε, δεν θα έχουμε πολύ χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικέ οι πληροφορίε που λαμβάνουμε από του εμπειρογνώμονε. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Μα μιλήσατε για μια σχέση, σύνδεση μεταξύ της μητρική άδεια και των μισθολογικών διαφορών. Τι πιστεύετε λοιπόν ότι θα ήταν απαραίτητο. Ίσως η διεξαγωγή μιας ανεξάρτητης έκθεσης, μελέτης. Να κάνουμε διαχωρισμό των γυναικών που ποτέ δεν ε, ήταν σε άδεια μετρότητα γιατί δεν έχουν παιδιά και εργάζονται και με τις γυναίκες που έχουν πάρει άδεια Αυτό το μυστολογικό χάσμα δηλαδή ξεκινάει από την πρώτη εγκυμοσύνη και μετά. Αυτό θα έδειχνει κατά πόσον οι γυναίκες που δεν έχουν παιδιά λαμβάνουν επίσης χαμηλότερους μισθούς. Σε περίπτωση, στην περίπτωση αυτή υπάρχει διακρατική μεταχείριση. Πρόκειται λοιπόν για τη διακρατική μεταχείριση ή πρόκειται για συνέπεια της μητρότητας. Καλό θα ήταν λοιπόν σε μία μελέτη να διαχωριστούν αυτές οι δύο ομάδες. Ένα λεπτό, λέει η Πρόεδρος σε κάθε μία από τις ομιλήτριες για να απαντήσουν. Ένα λεπτό για όλα. Ναι, ναι, ναι, πολύ λυπάμαι. Να διαλέξω ένα από τα ζητήματα που μου θέσατε ως ερωτήσεις. Νομίζω ότι η παρακολούθηση τα αναφέρατε πολύ μόνο. Οι επιθεωρήσεις εργασίας, ποιότητας, θα μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα στην πράξη. Το γεγονός ιδιαίτερος ότι πολλές γυναίκες που έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση δεν πάνε στο δικαστήριο. Αυτό θεωρώ ότι σχετίζεται και με τον φόβο της θυματοποίησης, τον οποίο αν θέλετε, Θα πρέπει να εστιαστούμε στην πρόληψη. Έχουμε πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις, γιατί είναι χρονοβόρα διαδικασία, ε, με υψηλό κόστος, δεν υπάρχει πρόβλεψη νομικής αρρωγής. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα έλλειψης νομικών διατάξεων. Υπάρχει από το 57 η σχετική πρόβλεψη της συνθήκης, η διάταξη της συνθήκης. Εδώ και πάρα πολύ καιρό η αρχή μισθολογικής ισότητας που θα πρέπει να ισχύει στα κράτη-μέλη. Νομίζω όμως ότι η εφαρμογή στην πράξη ανάλογα με το άτομο το οποίο θα πρέπει τελικά να στραφεί στα δικαστήρια όταν δεχτεί διακριτική μεταχείριση. Πιστεύω λοιπόν ότι το θέμα είναι πιο πολύ θέμα εφαρμογής. Αυτά πρόλαβα να σας απαντήσω. Λυπάμαι. Θα ήθελα να φερθώ στην ερώτηση για τη μερική απασχόληση, για το part-time και μπορώ ήδη να παρουσιάσω και να τονίσω αυτά που είπα πριν. Αν δούμε τι έγινε ανάμεσα στο 2006 και 2012 για τη διαφορά των αμοιβών για τους εργαζόμενους στο part-time, πέρασε από 8% διαφορά το 2006 στο 16% το 2012. Λοιπόν, αν θέλουμε πιο χαμηλά από το μέσο όρο γενικά, αλλά με μεγαλύτερη αύξηση. Τι κρύβεται πίσω από αυτό. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι περισσότεροι, λόγω της κρίσης, πολύ περισσότεροι άντρες έχουν ε, πάρει θέσεις part-time και στα part time η διαφορά του φίλου υπάρχει λόγω μεγαλύτερης παρουσίας των ανδρών. Άλλος λόγος, το part-time είναι και πλέον κατάλληλο για, πολλά, για ανθρώπους με πολλά προσόντα, ειδικά προσόντα. Μπορεί να είναι και θετικό αν θέλετε αυτό, όμως στο πέρασμα από των ανθρώπων με ειδικότητε μεγάλε προ το part-time μπορούμε να καταλήξουμε στι ίδιε ανισορροπίε που διαπιστώνουμε για τι άλλε επαγγελματικέ κατηγορίε στο full-time. Όπω υπενθύμιζα, όσο αυξάνεται η γνώση σε μια θέση εργασία, αυξάνεται και η διαφορά μεταξύ των φίλων. Αυτό ίσω δεν είναι λογικό. Αυτά τα στοιχεία, αυτά μα δείχνουν τα στοιχεία όμω. Άλλο στοιχείο όσον αφορά. Α, μάλιστα Εντάξει, αυτά είχα να πω για την ώρα. I would like to... Να απαντήσω στις ερωτήσεις της κυρίας Μορβάη από την Ουγγαρία. Ρωτήσατε γιατί τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν τα συστήματα αυτά σε ό,τι αφορά τα συστήματα αξιολόγηση και κατάταξης θέσεων απασχόληση. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν προβάλλεται επαρκώς στην οδηγία, εν συντομία μόνο αναφέρεται. Και επίσης πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη σε ότι τα συστήματα τα οποία φαίνονται τόσο αντικειμενικά σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι, συχνά μάλιστα, δεν είναι αντικειμενικά. Είναι πολύ πολύ στερεότυπα. Και αυτά τα στερεότυπα λοιπόν αποτρέπουν ε, τα κράτη-μέλη από το να είναι ουδέτερα, γιατί δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν προβλήματα ενδεχομένω στο σύστημα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορεί να διακινδυνεύσουν την αρχή της ίσης ε, αμοιβή. Μάλιστα. Εγώ να απαντήσω σε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση της κυρία Σόντροβα για την αποζημίωση για τις γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά τους. Δύο τρόποι υπάρχουν να το πετύχουμε αυτό. Συντάξεις ε, σε κάποιες περιπτώσεις προστίφονται ένσημα, για παράδειγμα. Αν οι γυναίκες έχουν αφιερώσει χρόνο για την αντροφή του παιδιού στο σπίτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως εδώ είναι το εξής το αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει οι γυναίκες να έχουν την ευκαιρία να επανέλθουν στην αγορά εργασίας σε τυπικές ε, μορφές ε, απασχόλησης. Αλλά εδώ το κράτος πρόνοιας θα πρέπει να παρέχει υπηρεσία, φύλαξη, βρεφονιπιακού σταθμού και η ανάγκη να ε, συμμετέχουν πιο πολύ οι άντρες, ο πατέρας. Δεύτερο θέμα για τις επιθεωρήσεις εργασίας. Οι επιθεωρήσεις εργασίας λειτουργούν, αλλά αυτό που καταδεικνύουν οι, έκθεση, οι εκθέσεις, για παράδειγμα η πρόσφατη έκθεση στην Πολωνία, είναι το εξής. Ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει διαμάχη μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ο εργαζομένος καν δεν θέλει να αναφέρει τίποτε, γιατί φοβάται για την θέση απασχόλησή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ όλου. Να ευχαριστήσω, λοιπόν, όλους ε, τους προσκεκλημένους. Να περάσουμε στο σημείο 5, έκθεση για το θέμα το οποίο μόλις συζητήσαμε. για την εφαρμογή της οδηγίας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η κυρία Σαμπόρφικα έχει το λόγο. Ah, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι η συζήτηση που διεξήχθη αποτελεί η αναπόσπαστο τμήμα της συζητήσεως που αφορά την έκθεσή μου. Έχουμε μπροστά μας ένα σχέδιο εκθέσεως που έχει στόχο να προτείνει λύσεις. Δηλαδή, πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη ισότητα των ευκαιριών και την ισότιμη αντιμετώπιση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία, το πρόβλημα αυτό απετέλεσε αντικείμενο πολλών εκθέσεων. Εδώ και μερικές εβδομάδες συζητήσαμε το ίδιο πρόβλημα στην έκθεση του συναδέλφου Μάρκ Ταραμπέλα. Μετά δέκα χρόνια εμπειρίας που απεκόμισα από τη θέση μου ως βουλευτής και ως μέλος της Επιτροπής αυτής προσπάθησα δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά να περιγράψω την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τους άνδρες και γυναίκες τις διαφορές όσον αφορά τους μισθούς και τις διακρίσεις στον τόπο εργασίας και απ' την άλλη έλαβα υπόψη επίσης τις θέσεις των συναδέλφων στο Κοινοβούλιο καθώς και τις θέσεις του Συμβουλίου. Προσπάθησα να προτείνω στην έκθεσή μου πράγματα ρεαλιστικά που να μπορούν να υιοθετηθούν στη ψηφοφορία. Πολλά στοιχεία ήδη αναφέρθηκα κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας. Θα έχετε δει την έκθεσή μου, θα την έχετε μπροστά σας, μεταφρασμένη στις γλώσσες, στις διάφορες. Είναι λοιπόν κάτι που προξενεί έκπληξη. Συζητούμε πάντα αυτό το πρόβλημα από το 1957 όπου εκεί υιοθετήθηκε η αρχή της μη διάκρισης στην συνθήκη της Ρώμης και υπάρχουν, υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο, πολλές αποφάσεις και όμως εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα προσυζήτηση. Θα ήθελα να σας πω ότι η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις αμοιβέ εξορισμού λαμβάνει υπόψη τρία χαρακτηριστικά. Όπως είναι η παιδεία, τομεακά χαρακτηριστικά, μέγεθος επιχειρήσεων Φερρυπίν και επίσης θεσμικά χαρακτηριστικά παραδείγματος χάρη ελάχιστη μισθή. που δεν καθορίζονται με νομικά ε, υποχρεωτικό τρόπο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, πρέπει να πούμε από την άλλη βέβαια ότι αυτή η διαφορά, όπως ανέφεραν και οι πυρογνώμονες, οφείλεται και στις θέσεις εργασίας σε μερική απασχόληση που έχουν διαδοθεί πάρα πολύ σε τομείς της υγείας, στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών, ε, στον τομέα καθαρισμού Φερρυπίν. Δημιουργείται λόγω της διαφοράς ε, και ανισορροπία και στον οικογενειακό χώρο και τον επαγγελματικό για τις γυναίκες. Συχνά οι γυναίκες αντιμετωπίζουν φτώχεια και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην εκπαίδευση των παιδιών και στις ε, γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά. Επηρεάζεται η εκπαίδευσή τους με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και διάκριση στον τομέα των συνταξιοδοτικών. Μας εκπλήσει το ότι αυξήθηκε η διαφορά των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυξάνεται η διαφορά όταν βγουν στη σύνταξη οι γυναίκες. Μέσος όρο είναι 39% η διαφορά. Στις χώρες, άλλες χώρες η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια. Η διαφορά είναι διπλάσια στη συντάξη μεταξύ ανδρών και γυναικών, εν συγκρίση με τη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν δούμε και την φτώχεια που επικρατεί όσον αφορά τις ηλικιωμένε γυναίκες, βλέπουμε ότι αυτή η διαφορά οδηγεί σε διακρίσεις και πρέπει να εξαλειφθεί. Τρία σημεία ακόμα θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, την έννοια της ίδιας εργασίας. Η έλλειψη ορισμού ή μιας εργασίας ίδιας αξίας ή να υπάρχουν στοιχεία αξιολόγησης ε, σαφή για τον καθορισμό ίδιας δουλειάς είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για να κινηθούμε προς μια αγορά εργασίας που θα είναι δίκαια, που θα βασίζεται στην ισότητα ανδρών και γυναικών και την ισότιμη αντιμετώπιση των δύο φύλων. Θα πρέπει να επιμείνουμε επί του ορισμού της ίδιας εργασίας ή μιας εργασίας με την ίδια αξία, αντίστοιχη αξία. Έχουμε την οδηγία του 2006, η οποία αναφέρει ότι υπάρχουν τέσσερα στοιχεία επί των οποίων προβασιστούμε γι' αυτό. Οι ικανότητες, η προσπάθεια, η ευθύνη, η υπευθυνότητα μάλλον και οι συνθήκες εργασίας. Άλλο στοιχείο, η διαφάνεια όσον αφορά τις αμοιβέ, τους μισθούς. Η θέσπιση μέτρων περί μισθολογικής διαφανείας επιτρέπει επίσης να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να δημιουργήσουμε μια αγορά εργασίας που θα βασίζεται στην ισότητα ανδρών και γυναίκων. Αν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, είναι δυσχερέστατο να στραφούμε προς τη δικαιοσύνη. Εάν δεν έχουμε ορισμό και διαφάνεια, δύσκολο οι γυναίκες να ε, υποβάλουν καταγγελίες και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Τέλος, πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Αναφερθήκαμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι η πρόσβαση στην δικαιοσύνη για τα θύματα διακρίσεων αποκλίνει κατά πολύ, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Θα ήθελα λοιπόν στην έκθεσή μας να υπογραμμίζουμε την ανάγκη νομικής αρρωγής, δωρεάν αρρωγής, νομικής που θα χορηγείται είτε από τους κρατικούς φορείς, τους υπεύθυνους για την ισότητα, είτε από τα συνδικάτα, είτε από μια μη κυβερνητική οργάνωση, θα πρέπει να βρούμε λύση στο Λουξεμβούργο. Γνωρίζω ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις γυναίκες παρέχεται δωρεάν. Είναι μια γυναίκα, ο... συγγνώμη, είναι μια χώρα που οι γυναίκες κέρδισαν τα περισσότερα και μπορούν να προσφεύγουν πιο εύκολα στη δικαιοσύνη. Αυτή η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι βασικό προαπαιτούμενο για την εφαρμογή των διατάξεων ε, περί δικαιοσύνης όσον αφορά τις αποζημιώσεις και για τις κυρώσεις. Η συνάδελφος αναφέρθηκε στις κυρώσεις. Θυμάμαι τη συζήτηση με θέμα την έκθεση της κυρίας Μπάουερ. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευθεί συνένεση όσον αφορά τις κυρώσεις, διότι θέλουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες από τη μια και από την άλλη πρέπει να σεβαστούμε και την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή της επικουρικότητας αναφέρεται πάντα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να βρούμε λύση αν προβλέπονται κυρώσεις όσον αφορά στη συμμε... όσον αφορά τις διαδικασίες σε δημόσιους διαγωνισμούς και ε, όσα, όσων τέτοιων διαδικασιών ε, εμπλέκουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σαν μια επιχείρηση το χάρη που ασκεί τις ε, τις διακρίσεις ενδιαφέρεται για πόρους που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ιδέες που θα μου δώσετε, διότι είναι πάρα πολύ ευρύ το πρόβλημα, είναι ευρέως διαδεδομένο και ελπίζω ότι υιοθετώντα την έκθεση μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση, από αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ η κυρία Γιέλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την πολύ καλή έκθεση της κυρίας Ζαμπόρσκα. Να συγχαρώ την κυρία Ζαμπόρσκα για αυτό γιατί υιοθετεί τις γραμμές που έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και εκφράζω τη στήριξή μου στα βασικά ζητήματα που είναι το αίτημα για αναθεώρηση της οδηγίας, αυτό είναι στο σημείο 20 των συστάσεων, είναι πολύ σημαντικό για μένα ε, σε αυτή τη νέα εποχή να το προσπαθήσουμε. Γίνεται μεγάλος λόγος για την κρίση, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να έχουμε νέους όρους μισθολογικής δικαιοσύνης. Και επίσης εκφράζω τη στήριξή μου στο θέμα των κυρώσεων. Βρήκατε ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να συμβάλλουμε. Να ακομίσουμε ευρωπαϊκή αξία. Και αυτό θα χρησιμεύσει και σε άλλες επιχειρήσεις για να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ποιο ε, κομμάτι της καταλαμβάνει ε, το μεγάλο θέμα της ισότητας. Επίσης, όλα αυτά που έχουν σχέση με τη μισθολογική διαφάνεια είναι πολύ σημαντικά και επιδέχονται πολλών βελτιώσεων, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν το λέω επειδή είναι της μόδας και δεν είμαι καταρχήν ε, θετική, διότι πολύ συχνά όλα αυτά τα θέματα με κάνουν επιφυλακτική γιατί θεωρώ ότι οι κυρώσεις και οι χρηματικές απειλές ουσιαστικά είναι βαρύδι ενώ αντίθετα θα έπρεπε να δίνουμε περισσότερα κίνητρα. Παρόλα αυτά σίγουρα πρέπει να ε, δείξουμε ποια κράτη-μέλη δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και σίγουρα στην Ευρώπη το θέμα των συντάξεων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Οι γυναίκες είναι φτωχές, οι φτωχές γυναίκες ούτως ή, οι γυναίκες ούτως άλλως ζουν περισσότερο και άρα οι φτωχές γυναίκες που δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στη σύνταξη δυσκολεύονται περισσότερο. Από την άλλη έχουμε την θηλυκοποίηση, να το πω έτσι, των ορισμένων επαγγελμάτων που ήταν καθαρά ανδρικά στο παρελθόν, αλλά λόγω κρίσης οι γυναίκες ε, τα ασκούν όλο και περισσότερο και υπάρχει επιδείνωση των συνθήκων, υπάρχει μισθολογική ανισότητα. Όλα αυτά τα προβλήματα οξύνονται και πρέπει να τα δούμε. Στο σημείο 26 όμως, στις συστάσεις λέτε ότι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μελέτη όπου θα συγκρίνει την κατάσταση των μητέρων με παιδιά και χωρίς. Ποιος είναι ο στόχος αυτών για αυτό το αίτημα. Με δεδομένη στις συνθήκες, τη μεγάλη αβεβαιότητα, την εργασιακή. Πολύ συχνά Έχουμε ε, μητέρες βεβαίως χωρίς παιδιά, μητέρες που δεν έχουν καν θέση στον εαυτό τους το ερώτημα γιατί είναι τόσο ηφαισιακή η κατάσταση και τόσο αβέβαιη η αγορά εργασίας που δεν έχουν τολμήσει να εξετάσουν το ενδεχόμενο του να κάνουν παιδιά. Πρέπει να έχουμε υπόψη όλη αυτή την αβεβαιότητα ε, που υπάρχει σε σχέση με τις γυναίκες και ειδικότερα όταν είναι ε, μητέρες ε, σε μονογονεϊκές οικογένειες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σοϊρόβα, παρακαλώ. Oui, merci. Je voudrais... Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο, την κυρία Άννα Ζαμπόρσκα, Και θα ήθελα να μιλήσω για αυτούς τους τρεις κλάδους, την αδικία, την αξιοπρέπεια των γυναικών και την αξιοπρέπεια στη μητρότητα. Οι γυναίκες είναι αυτές που τιμωρούν την κοινωνία αρνούμενες να κάνουν παιδιά. είναι η λογική τιμωρία, η λογική κύρωση όλης της κοινωνίας. Δυστυχώς, το ποσοστό γονιμότητας έχει καταβαραθρωθεί. Είναι απαραίτητη η οδηγία και ο κανονισμός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. η στήριξη ε, των γυναικών εκτιμάται καλύτερα και ο γονεϊκός του ρόλος εκτιμάται καλύτερα. Οι κυρώσεις ισχύουν για όλη την κοινωνία, για όλο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο οποίος υφίσταται τεράστιο πλήγμα από τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιούτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαμπόρσκα για την εξαιρετική της έκθεση. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεσή σας, άκουσα τους εμπειρογνώμονες, τους ειδικού. Πρέπει να πάρουμε την κοινή απόφαση να αναθεωρήσουμε αυτή την οδηγία. πρέπει να το δει και η Επιτροπή για τις κοινωνικές υποθέσεις. Εκεί εκπονούμε προτάσεις. Η μισθολογική ανισότητα ανδρών και γυναικών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να δίνουμε κοινό ορισμό στο, τις λέξεις αντίστοιχη εργασία ή εργασία αντίστοιχης αξίας. Να τονίσουμε τη διαφάνεια κατά τον υπολογισμό του μισθού και έτσι μόνο μειώνονται οι μισθολογικές ανισότητες ως προς το naming and shaming. Είναι χρήσιμη η υιοθέτηση αυτής της αρχής. Και ως προς τη μητρότητα Ελπίζω αυτά να μην περάσουν απαρατήρητα οι γυναίκες. Ε, γνωρίζουν πολλές διακρίσεις λόγω της μετρότητας. Όλοι μαζί ελπίζω θα είμαστε σε θέση να, κατα... εκπονήσουμε πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε όλους όσους παρενέβησαν. Καταχώρησα τις ερωτήσεις που ετέθησαν από την κυρία Γιάλα Σέντερ εξήγησα λίγο γιατί θα ήθελα να έχω δύο μελέτες, δύο τοποθετήσεις, διότι δείχνουν ότι αυτό το pay gap, η διαφορά, ξεκινά με την πρώτη, μετά την πρώτη γονική άδεια. Οι γυναίκες χωρίς παιδιά δεν έχουν διαφορά. Αν βάλετε μαζί τις άτεκνες γυναίκες και τις γυναίκες με παιδιά ίσως να έχουν ε, μεγαλύτερη ζημιά εις βάρος των γυναικών με τα παιδιά διότι το pay gap είναι υψηλότερο από το 16% που δείχνουν οι μελέτες και τα αποτελέσματα των μελετών μπορούν να δείξουν και τον αντίχτυπο της μητρότητας των γυναικών με παιδιά τι αντίκτυπο έχουν ε, οι διαφορές αυτές για την ευημερία της κοινωνίας. Για να έχουμε ένα σαφές αποτέλεσμα, να δούμε αν η μητρότητα πράγματι προξενεί τη διαφορά ή η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό, απλώς. Σας ευχαριστώ, πραγματικά σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας και χαίρομαι όλος ιδιαιτέρως, περιμένω τις τροπολογίες σας και περιμένω και τη συζήτηση. Θα, θα έχουμε μια συνεδρίαση για να συζητήσουμε και τις τροπολογίες και για να καθορίσουμε τις θέσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ζαμπόρσκα. Η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση είναι 15η Απριλίου το μεσημέρι. Θέλετε να μιλήσετε κι εσείς. Ναι. Ναι, θα ήθελα να πω κι εγώ το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. κυρίες. Θα είμαι σύντομη γιατί έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό έργο η κυρία Ζαμπόρσκα στο έργο της, στο, στην έκθεση της. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, ούτε θέλω να τοποποιήσω το περιεχόμενο. Υπήρχε το θέμα της εφαρμογής για την ίση μεταχείριση στον χώρο εργασίας, αλλά η συνάδελφος ε, Ζαμπόρσκα κατέδειξε ότι και το υφιστάμενο δίκαιο, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν κινείται πάντα προς την επιθυμητή κατεύθυνση με την ταχύτητα που θα θέλαμε. Καλό λοιπόν θα ήταν να υπάρχουν διατάξει για τη μητρότητα που να ε, καταδεικνύουν και τα πλανεκτήματα, τα οικονομικά πλεονεκτήματα, να ξέρουμε ποιο είναι το όφελο του να υπάρχει, του να φροντίζει η γυναίκα, τα παιδιά και την οικογένεια. Κάτι άλλο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για το γεγονός ότι δεν πληρώνεται για παράδειγμα η εργασία των γυναικών σε θέματα φύλαξης για να βελτιωθεί η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση περιλαμβάνεται και μία πρόταση, μία φράση ό,τι αφορά τα ποσοστά συντάξεων ε, για τις γυναίκες που είναι πιο χαμηλά. Θα πρέπει να υπάρχει εξίσωση των δικαιωμάτων, των συνταξιωτικών δικαιωμάτων. Και θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και το ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες οι μητέρες, χωρίς να υπάρχει διακριτική μεταχείριση η εργασία των γυναικών στην ε, οικογένεια. Δεν εκτιμάται αυτό επαρκώς σήμερα, παρά το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό συμβάλλει στην ευημερία του συνόλου. Και εδώ θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν σχετικοί δείκτες και να εξετάσουμε ποιοι είναι, ποιες είναι οι κατάλληλες μέθοδοι για την υπολογισμό του ρόλου αυτού. Και όλα αυτά να γίνονται με ουδέτερο τρόπο ως προς το φύλλο. Όντω λοιπόν υπάρχουν, διαφορά, υπάρχουν διαφορές στην ε, αμοιβή, στην αποζημίωση που προέρχονται από διακριτική μεταχείριση. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι κάνουμε ένα σωστό βήμα προς την κατάλληλη κατεύθυνση για την καλύτερη αναγνώριση των γυναικών. Δεν θα κάνω πολλές τροπολογίες όπως σας είπα, αλλά κάποιες ε, τροπολογίες θα ήθελα να σας, την... Ε, να σας εξηγήσω την ιδέα της εναρμόνισης για παράδειγμα. σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους. Στην πράξη, πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την κατάταξη και την αξιολόγηση, ύστερα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πρόταση που έγινε για την αντιστροφή του βάρους απόδειξης και ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών. Το θέμα των ένωμων μέσων, το θέμα των νομικών εγγύησεων που μπορούν να προβλέψουν οι εργαζόμενοι και οι εργαδότες. Αλλά δεν θα ήθελα να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της ε, συνολική μεταφορά του βάρου απόδειξη στον εργοδότη που δεν έχει κάνει ενδεχομένω ε, τίποτα το μεμπτό. Θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία και πιστεύω επίση ότι οι υποχρεώσει για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν θα πρέπει να είναι οι ίδιε απαραίτητα όπω αυτέ που βαρύνουν τι μεγάλε επιχειρήσει. Και ω προ ε, αυτό θα ήθελα να προτείνω μια. Ναι, θα θέλετε να Κλείνετε. Να ολοκληρώσετε, λέει η πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ολοκληρώνω. Δεν είναι επίση ε, σαφέ, πιστεύω, τι θα γίνει με την έρευνα για μητέρε ε, και για τι μητέρε, τι γυναίκε που δεν έχουν ε, παιδιά. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό το σημείο τη σημερινή διάταξη. Άλλο ένα έχουμε αλλά για προφανείς λόγους, επειδή πρέπει να τηρήσουμε και το χρόνο εργασίας των διερμηνέων, θα το αναβάλουμε το θέμα αυτό. Επρόκειτο για την οδηγία για την ε, γονική άδεια. Έχουμε αναθέσεις εξωτερική έρευνα αυτό το θέμα, αλλά επειδή θα μας ε, καταλήψουν οι διερμηνείς, θα παρακαλέσουμε να συνεχιστεί το θέμα αυτό στα αγγλικά. Και θα σας παρακαλέσω να συνεχίσετε λοιπόν στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ. Try to be brief, though uh, we are now turning to other directive and you must realize that there are many questions. Έχουμε πολλές ερωτήσεις από αυτήν την οδηγία. Μπορούμε να μόνο σε μερικά στοιχεία προσήγησα την οδηγία από πλευράς νομικών διατάξεων. Ενδιαφερόμουν όμως και για τον πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η οδηγία στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσω με συγκεκριμένες διατάξεις. Επεκτάθηκε η ελάχιστη διάρκεια της γονικής αδείας από τρει σε τέσσερι μήνες, σημαντικότερη αλλαγή. Από την ανάλυση μου είδα ότι έχουν εφαρμόσει όλες τις χώρες τη διάταξη Βέβαια ε, υπάρχει ποικιλομορφία διάρκειας. Οι περισσότερες χώρες παρέχουν γονική άδεια από 6 μέχρι 12 μήνες. Άλλη σημαντική διάταξη. Ένας μήνας θα πρέπει να είναι δικαίωμα ατομικό και μη μεταφερόμενο. Ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδέτερη από αυτού. Έπρεπε οι χώρες να έχουν κίνητρο να δώσουν ένα μήνα μόνο για τον πατέρα. Σύμφωνα με την ανάλυση που έκανα, από τις 18, οι 18 χώρες συμμορφώθηκαν. Και όπως βλέπετε είναι επικοινόμορφη αυτή ε, η, η ομάδα χωρών από διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κάποια σαφής υποδιέρεση που να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επόμενο σημαντικό είναι ότι το όριο ηλικία του παιδιού πρέπει να είναι μέχρι 8 ετών. Η γονική άδεια πρέπει να είναι διαθέσιμη μέχρι το παιδί να είναι 8 ετών. Ο λόγος για την θέσπιση της διάταξης ήταν η χρήση της γονικής αδείας να γίνει πλέον ευέλικτη. Όπως βλέπετε, από τις μόνο 6 χώρες έχουν συγκεκριμένο ρητό ε, όριο ηλικία που έχει καθοριστεί στα 8 έτη. Οι περισσότερες χώρες έχουν σταθερές συγκεκριμένη πρόβλεψη. Και ίσως η άδεια να χρησιμοποιηθεί με τη μία σε δύο τμήματα και για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Κυρίως σε χώρες που η άδεια είναι διαθέσιμη για δύο ή τρία χρόνια. Θα ήθελα ξανά να αναφερθώ εν συντομία στο θέμα των αμοιβών. Δεν αναφέρεται ρητά στις οδηγίες τι είδους εισοδηματική αποζημίωση συνοδεύει το δικαίωμα χρήσεως της αδείας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν διάφορα αποτελέσματα. Έχουμε γονική άδεια ανεφοποδοχών σε αρκετές χώρες, έχουμε κατακοποκοπήν πληρωμές, ένα μικρό ποσό κάθε μήνα, για 2, 3, 4 χρόνια σε κάποιες χώρες και έχουμε και κάποιες χώρες που είναι αρκετά γενναιόδορες όσον αφορά τις αμοιβέ, ακόμα και μετά στο επίπεδο 80 μέχρι 100% του μισθού. Πάω στο δεύτερο τμήμα της εκθέσεως, ποιες είναι οι κοινωνικές συνέπειες που επιφέρει η οδηγία. Πρώτη ερώτηση, ποιος χρησιμοποιεί την άδεια. Δεν θα σας εκπλήσει, περισσότερο οι γυναίκες χρησιμοποιούν την άδεια. Βλέπουμε εδώ ποσοστά ανδρών προς γυναίκες ανάλογα με τη διάρκεια της άδεια. Για συντομότερα χρονικά διαστήματα, περίπου μια μισή φορά περισσότερες γυναίκες μου από την άδεια. Όσον αφορά την άδεια που λαμβάνεται για πάνω από 12 μήνο, έχουμε 36 φορές περισσότερες γυναίκες από άνδρες. Άρα ε, είναι εκπληκτικό που οι γυναίκες ε, χρησιμοποιούν περισσότερο τη γονική άδεια. Αν δείτε πιο κοντά τον μέσο όρο των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δούμε το ποσοστό των διαθεσίμων ημερών είναι 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10% χρησιμοποιούν τις αδείες, 10% άνδρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν την άδεια αυτή. Αν δούμε στατιστικά στοιχεία για τους ε, άντρες που πρέπει τουλάχιστον μία μέρα άδεια, δεν χρησιμοποιούν όλο το δικαίωμά τους, τουλάχιστον μία εβδομάδα χρησιμοποιούν δύο εβδομάδες στην άδεια, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κρατών μελών και αν δούμε και τις χώρες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στη γονική άδεια βλέπουμε ότι τα συστήματά τους είναι πιο γενναιόδωρα από τις διατάξεις οδηγίας. Συνήθως πάνω από ένα μήνα, δύο-τρεις μήνες άδεια παίρνουν οι άνδρες. Οι που χρησιμοποιούν την άδεια ε, εισπράττουν και πληρωμή και πρέπει να είναι γενναιόδοροι αυτοί για να αντικαταστήσει την απώλεια εισοδήματο για τους άντρες αυτούς όταν χρησιμοποιούν τη γονική άδεια. Και μετά, αν δούμε γενικά τα αποτέλεσμα της οδηγίας, ίσως είναι έμεσα αν ήθελε ο νομοθέτη να βελτιώσει την ονοπία των φίλων όσον αφορά τη γυναίκα και οδηγία, αν ο νομοθέτη ήθελε να βοηθήσει τη συμφιλίωση οικογενειακή ζωή και εργασία, η πρόοδο είναι πολύ περιορισμένη. Μιλήσαμε για διακοπή των, ε, της διαφοράς, των διαφορών. Εδώ δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε τη διερμηνία. Θα συνεχίσετε στα αγγλικά. Καλό μεσημέρι.